Okay, colleagues. I still think these 2.30 starts. aren't really working. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήμουν σε αυτή την επιτροπή για πολλά χρόνια, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και καλώς ήρθατε λοιπόν στην κοινή μας συνεδρίαση με την, ε, την Επιτροπή Ανάπτυξης. Αρχίζεται πολύ νωρίς και πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ στις 6.30. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση. Περνάμε στο σημείο 26 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Δεν ξέρω ποιο σημείο είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. 15, 15. Έχουμε λοιπόν μια κοινή ανταλλαγή απόψεων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκθεση παρακολούθηση της προόδου προ την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμπρόεδρος μου, κυρία Βαλεάν, έχει πρόβλημα, είναι κολλημένη στην κίνηση και θα έρθει μόλις τα καταφέρει. Έχουμε τον κύριο Στόλα, δεν ξέρω αν λέω το όνομά σας σωστά, προσκεκλημένος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η δουλειά που κάνετε στην Eurostat και πώς ε, μετράτε την πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό διότι τον επόμενο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να παρουσιάσει την πρόοδο ε, σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης τόσο εντός όσο και εκτός της. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Ανάπτυξης συνεργάζονται μαζί σας από πέρυσι έτσι ώστε να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση της Ένωσης στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εστιάσαμε στην εξωτερική πολιτική μέχρι τώρα και πρέπει να εξασφαλίσουμε και συνοχή στην εσωτερική πολιτική με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Eurostat ε, δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση όπου παρουσιάζεται η πρόοδος ε, του κάθε κράτους μέλους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη ως προς τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσετε τους ε, στόχους, τι έχουμε καταφέρει, τι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και επίσης έχουμε προγραμματίσει μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας εν ώψη του 2019. Περιμένουμε έγκριση, γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε εγκαίρως τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν θα δώσω ευθύ, ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Στόιπερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, αντίστοιχης μονάδας τη Eurostat. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στόιπερ ονομάζομαι, επικεφαλής του τμήματος περιβάλλοντος στατιστικών και βιώσιμης ανάπτυξης της Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκομαι εδώ με την Κριστίν ε, Μάιερ, η οποία είναι αρμόδια για τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν την έκθεση παρακολούθησης για το 2018 σχετικά με την πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μπορώ να πω ήδη από τώρα ότι σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε την έκθεση νωρίτερα από ό,τι προγραμματίσαμε, πριν δηλαδή τον Ιούνιο, για να προλάβουμε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Να σας δώσω λοιπόν το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Γνωρίζετε ίσως ότι το θεματολόγιο το 2030 προβλέπει διάφορα επίπεδα παρακολούθησης σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό αναφέρεται ρητά στο θεματολόγιο του 2030. Θα σταθούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ένωσης μάλλον, αλλά είναι σημαντικό ίσως να σκεγγραφίσουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν το επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, παγκόσμιο επίπεδο, όπου η παρακολούθηση γίνεται ε, για 169 στόχους του θεματολογίου 2030 η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακας, αν θέλετε, οργανισμός, οι οποίοι συλλέγουν τα δεδομένα για την παρακολούθηση, η οποία λαμβάνει χώρα βασισμένη σε, 100, ε, σε 232 δείκτες. Είναι βασικοί ε, δείκτες ε, οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά. Το 40% όμως αυτών των 232 ε, δικτών αφορά δεδομένα από συγκεκριμένες χώρες. Ένα 30% ακόμα ε, αφορά δείκτες για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα και το τελευταίο 30% αφορά δείκτες για τους οποίους μέχρι τώρα δεν έχει συμφωνηθεί ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί. Έτσι εργαζόμαστε στα Ηνωμένα Έθνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Παρακολουθούμε την πρόοδο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο των ε, στόχων του ΟΗΕ. Εστιάζουμε σε βασικές πολιτικές της Ένωσης ε, με βάση για παράδειγμα την ανακοίνωση του 2016 για τα επόμενα βήματα προς μια βιώσιμη Ευρώπη. Η Eurostat και οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν κέριο ρόλο, αλλά και άλλοι φορείς της Ένωσης. Για την παρακολούθηση χρησιμοποιούμε το, την ομάδα δικτών ε, βιώσιμης ε, ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι δείκτες για τους οποίους έχουμε στατιστικά στοιχεία και ε, διεξάγουμε μια ετήσια αναθεώρηση έτσι ώστε να επικαιροποιούνται οι δείκτες αυτοί, διότι αλλάζουν ε, συχνά. Μετά υπάρχουν άλλα επίπεδα. Κάποιες χώρες έχουν δικές τους στρατηγικές για βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν δικούς τους εθνικούς δείκτες, οι οποίοι δεν είναι ταυτόσιμοι ούτε με τους ε, δείκτες των Ηνωμένων Αθηνών, ούτε με της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν δείκτες ε, παρακολούθησης, ε, θεματική τομής όπως για την ανεργία, για την απασχόληση, για την εκπαίδευση. Μετά γίνονται και κάποιες ασκήσεις, για παράδειγμα υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Bertelsmann, είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του για να μπορούμε να μετρήσουμε το πού βρισκόμαστε και το τι πρόοδο έχει σημειωθεί. Οι δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωση επιλέχθηκαν βασισμένοι σε δύο κύριου άξονε. Το επίπεδο πολιτική καταρχά, δηλαδή οι δείκτες πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τι πολιτικέ τη Ένωση και ε, η στατιστική τους αξία. Χρειάζεται δηλαδή μια ελάχιστη ποιότητα, οι δείκτες πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά κτλ επιλέξαμε το 2017 την αρχική ομάδα δικτών μετά από μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν τα κράτη-μέλη, διάφορες επιτροπές του Συμβουλίου, ένα φόρουμ χρηστών, πανεπιστημιακή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών αλλά και αρκετοί διεθνείς οργανισμοί. Η ομάδα των δικτών που δημιουργήσαμε βασισμένη στην διαβούλευση έχουν και την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Επιτροπής. Ε, το 2017 ε, έδωσαν και, εκείνη τη σύμφωνη γνώμη τους. Μετά υπήρχε και η ετήσια έκθεση ε, το 2017 επίσης που ήταν βασισμένη σε έξι δείκτες. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω για την αναθεώρηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και που θα αναφέρεται στην έκθεση του 2019 τα κύρια χαρακτηριστικά τη ομάδας ε, δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Υπάρχουν 100 διαφορετικοί δείκτες, ε, μοιρασμένοι εξίσου στου 17 ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 42 στόχοι χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, σκοπούς και στόχους, με απότερο στόχο να ενισχύσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 88 δείκτες επικαιροποιούνται σε αιτήσια βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παρακολούθηση. Τα δύο τρίτα των δεικτών προέρχονται από επίσημα στατιστικά στοιχεία και ε, το υπόλοιπο ένα τρίτο από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, για τους περιβαλλοντικούς δείκτες, ΟΣΑ ε, και άλλες ε, πηγές. 55 από τους 100 είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους και τους δείκτες των Ηνωμένων Εθνών και 28 ε, δείκτες είναι ευθυγραμμισμένοι με τις ευρωπαϊκές πολιτικές όπως Ευρώπη 2020, τις προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τον ε, πίνακα επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου για να σας παρουσιάσει την έκθεση αναλυτικότερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω το, τη δεσμέτρων παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο, διότι για να φτάσουμε ε, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ε, χρήστες στο ευρύ κοινό, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικές μεθόδους. Όλα αυτά θα τα βρείτε στον ιστότοπο της Eurostat. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορες εκθέσεις και θα σας παραπέμψω στη συνέχεια σε αυτά. Λοιπόν, Αναφέρθηκα ήδη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους Υπάρχει ένας κατάλογος από δείκτες. Ο Άντων ήδη σας εξήγησε εν συντομία πώς ε, λειτουργούν αυτοί. Αν πάτε λοιπόν στον ιστότοπό μας θα δείτε για τον κάθε στόχο βιώσιμης ανάπτυξης ε, τους δείκτες ε, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την αξιολόγηση. Βλέπουμε στα δεξιά για παράδειγμα εκπαίδευση, τους δείκτες για την ποιοτική εκπαίδευση. Θα δείτε επίση ότι για ορισμένου στόχους υπάρχουν ήδη κάποια νούμερα πρέπει να πιάσουμε. Για παράδειγμα για την εκπαίδευση έχουμε το πλαίσιο παρακολούθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάρχουν οι κύριοι δείκτες, η ομάδα δικτών που έχουν ε, καθορίσει τα κράτη-μέλη και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους επίσης. Όπου βλέπετε αυτόν τον, αυτό το σύμβολο που είναι σαν στόχος ε, υπάρχουν ε, ελλείψεις στην αξιολόγηση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον διαχωρισμό, Εάν υπάρχει ένας ε, στόχος, ε, μπορούμε να τον μετρήσουμε σύμφωνα ε, με την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Υπάρχει δηλαδή καλή πρόοδος, το πράσινο βέλος που δείχνει προς τα πάνω, μπορεί να υπάρχει μέτρια πρόοδος, είναι το διαγώνιο βέλος, το οποίο δεν υπάρχει σε, στο συγκεκριμένο στόχο βιώσιμη ανάπτυξη, στην ποιοτική εκπαίδευση δηλαδή που βλέπετε στη διαφάνεια. Ε, ανεπαρκής πρόοδος, δηλαδή υπάρχει πρόοδο, αλλά δεν αρκεί για να φτάσουμε το στόχο αυτό ή επίση μπορούμε να έχουμε μια απόκληση από του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί βλέπετε ένα κόκκινο βέλο που δείχνει προ τα κάτω. Εάν δεν υπάρχει στόχο, τότε αξιολογούμε τι τάσεις προ τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν επίσης και διάφορες κατηγορίες ε, οι οποίες ε, αφορούν την πρόοδο από αρκετή ως μέτρια αλλά και την απόκληση, από μέτρη απόκληση ως και μεγάλη απόκληση. Τέσσερις λοιπόν κατηγορίες ε, που αφορούν τους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται. για κάθε στόχο βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται λοιπόν αυτή η αξιολόγηση, λαμβάνοντα υπόψη όλου του δείκτε και μετά καταλήγουμε σε μια συνολική αξιολόγηση, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Οι καλύτερε επιδόσει αφορούν του ε, στόχου 3, ε, υγεία, 4 ε, ποιοτική εκπαίδευση και 7 ενέργεια. Στα αριστερά σας θα δείτε ότι ο στόχος 10, δηλαδή μείωση της, των ανισοτήτων, έχει ελλείψεις. Δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο και μάλιστα παρατηρούμε αντίθετη τάση, επιδείνωση δηλαδή ε, της κατάστασης τα τελευταία χρόνια. Για του τέσσερι στόχου βιώσιμη ανάπτυξη που βρίσκονται κάτω, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τι τάσει, διότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογήσουμε του δείκτε και τις τάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ε, υπάρχουν λιγότερο από 75% ε, στοιχεία δεν μπορούμε να κάνουμε την αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αυτά λοιπόν ως προς ε, τους ε, δείκτες. Υπάρχει η έκθεση παρακολούθησης των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που θα έχετε λάβει όλοι ελπίζω. Το βιβλιαράκι αυτό στο οποίο υπάρχει μία λεπτομερής ανάλυση όλων των δικτών και παρουσίαση επίσης της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε. Υπάρχουν και διάφορα φυλάδια, αυτό το φυλάδιο το οποίο είναι πιο εύκολο στη χρήση του, δίνει μια συνολική εικόνα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν και νέα προϊόντα. Φέτος είχαμε μια νέα δημοσίευση και θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους να πάτε στον ιστότοπο μας και να το δείτε με τα μάτια σας, διότι ε, είναι αρκετά διαδραστική σωστό, σωστό μπορείτε οι ίδιοι να μαντέψετε την πρόοδο, μπορείτε να ε, χρησιμοποιήσετε διάφορα οπτικοακουστικά στοιχεία. Είναι αρκετά ελκυστικό σωστό τόπος για τους νεότερους χρήστες. Ε, έχει και στοιχεία παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Θα ξαναδώσω το λόγο στο συνάδελφό μου. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της παρουσίασης. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται μία ε, ακόμα αναθεώρηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο επίκαιροι και να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα στις ε, πρωτοβουλίες πολιτικής. Για παράδειγμα, οι δείκτες του κοινωνικού πίνακα του πίνακα κοινωνικών επιδόσεων είναι ένας από αυτούς τους τρόπους που χρησιμοποίησαμε και στους οποίους βασιστήκαμε. Στόχος μας είναι οι στόχοι να συνδέονται περισσότερο με την πολιτική, να αυξηθούν οι ε, δείκτες ποιότητας, αλλά και ε, να κρατήσουμε το ανώτατο όριο των έξι δικτών αλλά, ε, αναστόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, Υπάρχει άλλος ένας κατάλογος ε, με τις εκκρεμότητες, δηλαδή με τους στόχους που είναι καλή αλλά όχι αρκετά καλοί, οπότε είναι σε αναμονή και όλη αυτή η αναθεώρηση είναι αποτέλεσμα μιας ευρείας ε, διαδικασίας διαβούλευσης όπου ε, είχαμε την συνεισφορά διαφόρων φορέων, της πλατφόρμας για τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης, την Multi-Stakeholder Platform. Η αναθεώρηση των δικτών θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2018. Στις 23 Νοεμβρίου, θα, ε, την Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται, θα συναντηθούμε με τους ε, επικεφαλείς ε, των ετοιμάτων γενικών διευθύνσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον μόνο τρεις είναι οι δείκτες που θα αλλάξουν για φέτος. Υπάρχει αναθεώρηση το, της ομάδας των εδικτών και σε εμά και στα Ηνωμένα Έθνη. σε συνδυασμό με τις νέες πολιτικές με τον ορίζοντα 2020, τον οποίο θα αντικαταστήσει ένα νέο πρόγραμμα. Αναμένουμε λοιπόν να γίνει μια μεγάλη κλίμακα αναθεώρηση μετά το, για μετά το 2020. Θα δημοσιεύσουμε λοιπόν αυτήν τη νέα ομάδα δικτών που θα μοιάζουν πολύ με τους εφιστάμενους στις αρχές Ιανουαρίου και έπειτα θα συντάξουμε μια έκθεση την οποία ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε πριν το τέλος Ιουνίου 2019 έτσι ώστε δηλαδή να είμαστε, ε, να προλάβουμε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω να θέσω κι εγώ μερικές ε, ερωτήσεις και υπάρχουν και συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Θα ήθελα να γνωρίσω πώς συνεργαστήκατε με την Επιτροπή. Εσείς μας δείξατε συγκεκριμένες τάσεις, αλλά δεν αναφερθήκατε στα πολιτικά συμπεράσματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι ανισότητες φαίνεται να αυξάνονται. Φαίνεται ότι να μην υπάρχει καμία βελτίωση στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Περιμένουμε από από την Επιτροπή μέχρι το Δεκέμβριο να μας ε, υποβάλει ένα έγγραφο σε ό,τι αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό. Το ερώτημά μου είναι τι τις κάνετε αυτές τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές θέτουμε ορισμένου στόχους και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Μίλησα με την ε, κυρία Χάσελα και είπαμε ότι θα πρέπει να ε, παρακολουθούμε αυτά τα κοινά συμπεράσματα. Γίνεται, υπάρχει ένας μηχανισμός ε, αξιολόγησης μεταξύ ίσων ή δίνονται πληροφορίες μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή κρίνεται κατά πόσον κάθε μεμονωμένη χώρα επιτελεί κάποια πρόοδο. Γίνεται κάποια ανάλυση των δεδομένων. Βλέπετε στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς κινείται. Αυτό που είπατε είναι ότι υπάρχει έλλειψη μίας ενιαίας μεθοδολογίας ε, για τα κράτη-μέλη. Βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να αλλάξουν ε, οι μεθοδολογίες. Μία ακόμα ερώτηση από μένα. Έχετε αυτό το μηχανισμό αλληλεπίδρασης για, τις, ε, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ακόμα και οι νέοι άνθρωποι μιλάνε για το θέμα των βιώσιμων στόχων. Κάνετε κάτι σε συνεργασία με ορισμένους ε, φορείς ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες ενδεχομένως που προωθούνται σε σχολεία ή σε οργανώσεις. Αυτές είναι οι δικές μου ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια ερώτηση να κάνουν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Δίχως άλλο θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για τη δουλειά που φανταζόμαστε ότι θα κάνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι αυτοί που αποφασίζουν τις πολιτικές, η Επιτροπή, η ΟΚΕ, το Κοινοβούλιο, θα προσθέσουν μερικές ποιοτικές τυχές στο όλο θέμα. Αναφερθήκατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά των νέων. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα, μια ολόκληρη θεωρία ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Χθε κιόλα μια ομάδα παιδιών επισκέφθηκε το σχολείο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα τα παιδιά είπαν ότι είναι τρομοκρατημένα με αυτό που ενδεχομένω θα συμβεί στο πλανήτη. Το θέμα είναι αυτοί που αποφασίζουν το μέλλον, που αποφασίζουν τις πολιτικές, τι θα κάνουν. Όταν ήμασταν μικροί, κάναμε οικονομία στο νερό κλείναμε τις βρύσες, ε, ε, δεν πετάγαμε σκουπίδια. Ε, τώρα είναι σειρά άλλων. Θέλουμε να, δούμε τι ακριβώς κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα είδος συμμετοχικής διαδικασίας. η οποία δίνει ελπίδες και δίνει μία διασφάλιση ότι οι υπεύθυνοι κάνουν κάτι. Πώς θα γίνει αυτό μια ζωντανή διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα και έξω από αυτή την ε, αίθουσα. Ναι, μίλησα με νεαρούς ανθρώπους και μου είπαν ότι προβληματίζονται για το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Ήταν νεαρά παιδιά από την Πολωνία, από την ε, Σλοβενία Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει το ενδεχόμενο από αυτή τη βάση δεδομένων να δημιουργηθεί ένα δυναμικό αφήγημα. Ενδεχομένως υπάρχουν αποφάσεις που μας οδηγούν στο επόμενο βήμα και μας δίνουν περισσότερες ευκαιρίες εάν ολοκληρώσουμε την υπάρχουσα διαδικασία. Να υπάρξει δηλαδή μια καλύτερη ε, ρύθμιση, το Horizon Europe κτλ. Είμαι σίγουρη ότι θα πάρουν περισσότερο, ε, μέρος περισσότεροι άνθρωποι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλλατε και για την τόσο χρήσιμη αυτή έκθεση. Από την απαρχή των βιώσιμων στόχων επιμείναμε σε ό,τι αφορά την ανάγκη να παρακολουθήσουμε την πρόοδο στις διάφορες χώρες μέλη και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το θέμα είναι ότι η δουλειά που κάνετε πραγματικά βοηθάει, αλλά παράλληλα βλέπω ότι υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο πρώτος πρώτο όριο είναι η εφαρμογή όλων αυτών. Όταν βλέπω τις εκθέσεις ε, και βλέπω ότι γίνεται μία μέτρηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκέφτομαι ότι ενδεχομένως θα, έπρεπε να έχουμε να θεωρήσει αυτούς τους στόχους για να περάσουν να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτή ακριβώς τη συζήτηση είχαμε την Επιτροπή όταν μιλήσαμε για θέματα βιωσιμότητας. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο για μας αν στην έκθεση, αν είναι δυνατόν στην επόμενη επόμενη της έκδοση όχι μόνο να κάνουμε μία αξιολόγηση για την πρόοδο ή την ε, οπισθοχώρηση μερικών στόχων. Αν θα ήταν δυνατόν, έλεγα, να μετρήσουμε, να κάνουμε μετρήσεις ε, με μία αναφορά στην επίτευξη του στόχου. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα έχουμε ενδείξει για το αν να προοδεύουμε ή όχι. Θα ήταν δυνατόν στην έκθεσή σας να μας δώσετε μία ιδέα του πόσο απέχουμε από την επίτευξη του στόχου, γιατί νομίζω ότι και αυτό θα ήταν χρήσιμο. Διαπιστώνω ότι στις ε, διαφάνειες υπήρχε μία ε, που ε, αφορούσε, τον στόχο 10 που βρισκόμαστε πίσω σε ό,τι αφορά άλλα θέματα έχει επιτευχθεί πρόοδος. Ορισμένες περιπτώσεις σταθερή πρόοδος αν μία από τις πιο σημαντικές πτυχές του νέου θεματολογίου δεν είναι η παγκοσμιότητα αλλά το γεγονός ότι διασυνδέονται όλοι οι στόχοι μεταξύ τους νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένας τρόπος για να το τονίσουμε αυτό. Για να πούμε ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αν προοδεύουμε σε ό,τι αφορά ένα στόχο, προοδεύουμε παντού. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι διάφοροι στόχοι. Και πως η πρόοδος ε, σε ό,τι αφορά τον ένα στόχο δεν σημαίνει πρόεδρο, πρόοδο και τους άλλους αν παραμένουν ως είχαν. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να δείξω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια. Νομίζω ότι ήδη υπόθηκε αυτό. Είμαστε πολύ λίγοι εδώ. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε η δουλειά που κάνουμε σε ό,τι αφορά το θέμα των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης να γίνει μια συζήτηση ε, κατεστημένη, μια συζήτηση mainstream, να δούμε ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης και δεν θέλω να φανταστώ ότι μόνο έξι από εμά ενδιαφέρονται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι στην επόμενη συζήτηση θα παρίστανται περισσότεροι συνάδελφοι για να συζητήσουν τα σημαντικά αυτά θέματα. Τελευταίο σημείο, στην επόμενη έκθεση θα μπορούσατε να έχετε και μία αξιολόγηση του πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν και τις τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Βαλεάν ζήτησε το λόγο. Καλησπέρα σας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και εμείς ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος στηρίζουμε αυτά τα θέματα και έχουμε συμφωνήσει ήδη με πολλά από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Και πραγματικά είναι πολύ απογοητευτικό να αφιερώνουμε τόσο τεράστιο ε, μέρος των δραστηριοτήτων μας σε θέματα που έχουν πολύ χλωμή εξέλιξη. Όχι επειδή δεν έχουμε αποτελέσματα στις πολιτικές μας, αλλά λόγω της ε, εφαρμογής. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τόσες πολιτικές για να στηρίξουμε το πρόγραμμά μας για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά τι γίνεται με την εφαρμογή των μέτρων. Μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα. Γιατί εκεί είναι που χάνουμε, εκεί χωλαίνει η διαδικασία. Είδε μη, ε, θα μιλούμε στον κόσμο, όπω είπε η κυρία Χάουταλα, ε, όπως είπαν η Λίντα Μακάβαν, μιλούμε στον κόσμο και ο κόσμος φοβάται για, το πεπρωμένο του πλανήτη. Και εμείς μπορούμε να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ΑΒΓ νομοθεσία για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, για να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ωραία, αλλά αυτά είναι στη θεωρία. Πού είναι όμως η, η δράση, τα έργα, η εφαρμογή που πρέπει να γίνει σε επίπεδο κρατών μέλων. Η κλιματική βασικές δράσεις δεν μπορούν να καταμετρηθούν από ό,τι φαίνεται στη μελέτη. Γιατί αυτό το μήνυμα θα στείλουμε στο Κατοβίτσε στην διάσκεψη των μερών, ότι δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε την κλιματική μας δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι απλώς περιοριζόμαστε στα λόγια. Αλλά πού είναι η δράση, πού είναι τα έργα, πού είναι οι αποδείξεις. Νομίζω ότι έχουμε αρκετού δείκτες για να καταμετρήσουμε και τις κλιματικές δράσεις μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω όλους τους δείκτες, το. Πώς λοιπόν δεν μπορέσετε να καταμετρήσετε την κλιματική μας δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και για το καθαρό είδωρ και την αποχέτευση που είναι άλλος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης, πώς δεν μπορούμε να τα καταμετρήσουμε αυτά στα κράτη-μέλη. Είναι απίστευτο. Καθαρό νερό και αποχέτευση. Είναι δυνατό να μην μπορούμε να τα καταμετρήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Ακούσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση και εφαρμογή νομοθεσίας, για την ποιότητα του νερού. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αξιολόγηση για την ποιότητα του νερού. Πώς δεν μπορεί ε, να κάνει μετρήσεις λοιπόν για να δούμε κατά πόσο υλοποιούμε και σε τι βαθμό το σχετικό στόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλώς εκφράζω την απογοήτευσή μου, γιατί έχουμε αφιερώσει τόσο χρόνο και τέτοια προσπάθεια για πολλά θέματα ε, για τα οποία περιμέναμε πρόοδο, αλλά δυστυχώς πρόοδο δεν βλέπουμε. Και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό, γιατί είδαμε ότι έγινε ισμάτιν όλη αυτή η προσπάθεια. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ τη κλιματική αλλαγή την καταμετρούμε. Έχουμε τους στόχους μας για το 2020, για το 2030 και καταμετρούμε την πρόοδο ε, που υλοποιούμε και για το καθαρό νερό. Ε, βλέπουμε σε τι επίπεδα φτάνει η ποιότητα του νερού και έχουμε πολύ αυστηρά πρότυπα και προδιαγραφές για την ποιότητα του νερού. Βέβαια, αν δεν συγκεντρώνουμε αυτά τα στοιχεία, πώς θα το εξηγήσουμε στο Κατοβίτσε, στη διάσκεψη των μερών, και να πούμε ότι δεν έχουμε στοιχεία. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά κατά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από μια πιο στατιστική σκοπιά και μετά οι συνάδελφοι θα ασχοληθούν με τα πιο ακαθόδη ζητήματα της πολιτικής. Να ξεκινήσω καταρχήν με το ρόλο της Eurostat σε αυτή τη διαδικασία. Και στο, στο, στα Ηνωμένα Έθνη το ίδιο συμβαίνει ζήτησαν από τους στατιστικολόγους να κάνουν αυτή την παρακολούθηση ε, και να δημιουργήσουν το σχέδιο, το πλαίσιο της παρακολούθησης. Και αυτό είναι ουδέτερο. Εξετάζουν την ποιότητα των στοιχείων, αλλά δεν εμπλέκονται οι στατιστικολόγοι σε πολιτικά ζητήματα. Καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία. Καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη ποιότητα των δεδομένων τους στόχους πολιτικής δεν τους εφευρίσκουμε εμείς, τους ε, παίρνουμε έτοιμους από άλλους. Δεν είναι δικός μας ο ρόλος να φτιάξουμε την πολιτική και στο κείμενο κάνουμε την στατιστική περιγραφή. Τα πιο πολιτικά κείμενα για σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες προέρχονται από τις γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με τις πολιτικές. Εμείς απλώς τις περιλαμβάνουμε στη δική μας δουλειά. Και στη βάση δεδομένων θα βρείτε πληροφορίες για τα κράτη-μέλη και οι περισσότεροι δείκτες ε, ταξινομούνται και ανακράτως μέλος. Αλλά δεν βάζουμε ε, πράσινα ή κόκκινα βέλη ε, χαρακτηρίζοντας τα κράτη-μέλη, γιατί αν το κάναμε δεν νομίζω να ικανοποιούσαμε τα κράτη-μέλη και δεν είναι ρόλος μας αυτός να κατηγορήσουμε. Και εδώ το κλειδί βρίσκεται στην ερμηνεία. Και δεν ξέρουμε γιατί μια χώρα ε, θα μπορούσε να έχει πράσινο ή κόκκινο βελάκι αν δεν έχουμε τις εξηγήσει. και χωρίς εξηγήσει ε, δεν θα ήμασταν δίκαιοι. Σε ό,τι αφορά την προώθηση, φέτος για πρώτη φορά είχαμε και ψηφιακή ε, δημοσίευση για να φτάσουμε και στους νέους. Μέχρι στιγμής εκεί έχουμε φτάσει, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Αλλά δεν έχουμε σημαντικό μεγαλεπίβολες πρωτοβουλίε. Εμείς είμαστε στατιστικό γραφείο, παράγουμε στοιχεία, δεδομένα, τα δημοσιεύουμε όπως μπορούμε και βλέπετε ε, από το πακέτο, από τη δέσμη μέτρων υπάρχουν διάφοροι μορφοί διάδοση αυτών των στοιχείων. Ρωτήσατε αν μπορούμε να πούμε πόσο απέχουμε από την υλοποίηση του στόχου. Ποια είναι η απόσταση που μας χωρίζει από ένα στόχο. Αυτό γίνεται μόνο όταν έχουμε στόχο πολιτικής. Αν δεν έχουμε τέτοιο στόχο πολιτικής, ε, ε, δεν μπορούμε εμείς στο στατιστικό γραφείο να κάνουμε δήλωση για το πόσο απέχουμε από την υλοποίηση του στόχου. Αυτό το κάνουν οι γενικές διευθύνσεις που αφορούν, ασχολούνται με τις πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε, αλληλεπιδράσεις ε, με τρίτες χώρες, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και το σκεφτόμαστε. Το θέμα το, της κλιματικής δράσης. Εσείς αναφερθήκατε στην συνολική εικόνα και έχουμε τέσσερις τομείς που έχουμε και το ε, νερό και το κλίμα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μία ε, αθεριστική παρουσίαση, συγκεντρωτική. Ίσως για την κλιματική δράση θα μπορούσαμε να το κάνουμε το θέμα είναι ότι οι δείκτες που επιλέξαμε δεν μας επέτρεψε μια τέτοια προσέγγιση. Φέτος όμως θα το κάνουμε. Και αυτή η αθρηστική αξιολόγηση είναι ουσιαστικά ένας απλός μέσος όρος όλων των επιλεγμένων δικτών και είναι ένα επικοινωνιακό μέσο ώστε να μπορεί να αποκτήσει κάποιο μια γενική επισκόπηση. Πάντως οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι είναι υπεραπλουστευμένη αυτή η μέθοδος. Οπότε πάντα α, έχουμε το δίλημα θέλουμε να φτάσουμε λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό θα μας ε, περιορίσει σε μια απλή επισκόπηση. Οπότε οι εμπειρογνώμονες που θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο θα μας ε, κατηγορήσουν. Αν δώσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο θα μας κατηγορήσουν αυτοί που θέλουν γενική επισκόπηση. Για το νερό δεν είχαμε αρκετούς δείκτες ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και συγκεντρωτικά στοιχεία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και λίγα λόγια λοιπόν για το ευρύτερο πλαίσιο. Όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα πρωτοπόρος στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι αγκυροβολημένη η βιώσιμη ανάπτυξη στις συνθήκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει κέριο ρόλο στην ανάπτυξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κοινή ευθύνη όλων μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ε, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εφαρμόζει μαζί με τα κράτη-μέλη ε, το θεματολόγιο αυτό σε εθνικό, περιφερειακό και ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχει κάνει κάποια βήματα τα οποία αφορούν την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καταρχάς ευθυγραμμίζοντας τους στην ενωσιακή πολιτική, και επίσης ε, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα πολιτικής μετά το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αυτή τη στιγμή καταρτίζει ένα έγγραφο προβληματισμού για το, την εποχή μετά το 2020 και την εξέλιξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένης μάλιστα της Συμφωνίας του Παρισιού. Και να τονίσω εδώ ότι αυτό το όραμα είναι κυρίως πολιτικό. Ε, και στόχο έχει να τονώσει την ε, συζήτηση, να δώσει ιδέες και προβληματισμό. Είναι κομμάτι της ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη ευρωεκλογών, αλλά και πέρα από αυτές, μετά από αυτές. Είναι και κάτι το οποίο θα απασχολήσει την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε λοιπόν ε, στο τέλος του 2018 να εγκριθεί το έγγραφο προβληματισμού. Αν εσείς ε, θέλετε κάποια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, ε, καλό θα ήταν να δημοσιευθεί πριν το τέλος της θητείας. Αυτά λοιπόν και να σας πω ότι προσβλέπουμε στην συνέχιση της καλής μας συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ναι, καταλαβαίνω τα στατιστικά στοιχεία και τους στατιστικολόγους και αυτά που λένε, όμως ε, αυτό που δεν καταλαβαίνω πολύ καλά είναι το ότι δεν φαίνονται οι τάσεις των κρατών μελών, διότι αυτό δεν αρέσει στα κράτη-μέλη. Έχουμε δείξει τάσεις για το κάπνισμα, ε, για διάφορα άλλα πράγματα στην Eurostat και νομίζω πως ε, το θέμα εδώ είναι να μην έχουμε την απέτηση από τους στατιστικολόγους να μας εξηγούν το γιατί, αλλά να ε, συλλέγουν δεδομένα και να τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσουν ερωτήσεις από τους πολίτες. Ε, να ρωτήσουν δηλαδή οι πολίτες γιατί δεν πιάνουμε τους στόχους, γιατί γυρίζουμε πίσω, γιατί δεν πάμε μπροστά. Ο σκοπός των, ε, της συλλογής δεδομένων δεν είναι να δείξουμε ότι όλα πάνε κατευχήν, ο, ακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα. Το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όλα τα κρατημέλη, κάθε ένα από αυτά, υπέγραψαν το 2015 στα Ηνωμένα Έθνη εθελοντικά, από μόνα τους. Έχουν συμφωνήσει σε αυτά. Και να σας πω ότι πηγαίνω πολύ συχνά σε χώρες της Αφρικής και συναντιέμαι με υπουργούς, με ε, μέλη της κυβέρνησης και πολλοί ε, από αυτούς παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία, παρακολουθούν τις εξελίξεις και δεν ε, είναι δυνατόν εμείς οι ίδιοι να μην μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ελπίζω λοιπόν να σημειωθεί πρόοδος. μέχρι και στη θάλασσα, σε υποθαλάσσιο επίπεδο, ξέρουμε τη βιωσιμότητα των ειδών το θαλάσσιο ειδών. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να μετρούμε την πρόοδο στις κλιματικής ε, δράσης. Όπως είπε και η κυρία Βαλεάν, ε, μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδο προς τους ε, στόχους για το 2020. Εντάξει, ίσως διαφέρουν λίγο οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, όμως ήλπιζα οι στόχοι να είναι ξεκάθαροι. Και να πω κάτι στον Γενικό Γραμματέα το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και βλέπω πως καθυστερούν κάπως, ε, κύριε Γενική Γραμματέα, ε, τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2015 πήγε ο Επίτροπος στη Νέα Υόρκη και τώρα έχουμε 2019 σχεδόν. Και τι κάνουμε, έχουμε ένα έγγραφο προβληματισμού που προετοιμάζουμε. Αυτό είναι το πολιτικό όραμα μου θυμίζει λίγο την πολιτική δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για το μέλλον της χώρας, δηλαδή πολύ φανφάρα και περιεχόμενο μηδέν. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή για το Κοινοβούλιο, αλλά ελπίζω να δω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνητρο, να δω να κινούνται τα πράγματα προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, διότι χρειάζεται να δείξουμε τον ε, ηγετικό μας χαρακτήρα στο διεθνές ε, προσκήνιο, στην ε, ΚΟΠ, αν θέλουμε να μας ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ελπίζω λοιπόν να συνειδητοποιήσετε την επίγουσα κατάσταση και τον επίγοντα χαρακτήρα ε, Τη έκθεση αυτή και να προχωρήσετε. Θα σταματήσω όμως εδώ, διότι να... πρέπει να αφήσουμε και την κυρία Βαλεάν να μιλήσει. Να πω και εγώ δύο λόγια στήριξη αυτών που είπατε. Βλέπω τους δείκτες που έχω μπροστά μου. Και δεν βλέπω κάποιον δείκτη που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους τομείς ε, στους οποίους αναφερθήκατε, τους τομείς που είναι δύσκολο να μετρήσουμε. Δεν νομίζω πως ε, κάνουμε πυρηνική φυσική εδώ. Λέτε πως δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τα κρατημέλη, να τα φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτό όμως είναι ε, δυσάρεστο και αν έβγαζα συμπεράσματα τόσο εύκολα θα έλεγα ότι όποιος διαβάσει την έκθεση θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα ότι δεν ε, συμπεριλαμβάνονται δεδομένα εδώ διότι θα ε, πέσει η υπόλοιψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα δούμε ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ άσχημα στην αποχέτευση, στο καθαρό ε, νερό, στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε το. Πρέπει να ασχοληθούμε με τους δείκτες και να τους συνοδεύσουμε με δεδομένα, με στατιστικά στοιχεία. εάν τα αποτελέσματα είναι τόσο άσχημα και οι επιδόσεις μας τόσο χαμηλές, πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι οι πολίτες ε, θα το καταλάβουν, διότι θα ε, γυρίσουμε ε, ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτά από μένα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Πρόεδρό της που ήρθαν και προσβλέπουμε στην δημοσίευση της έκθεσης. Μάλιστα. Ε, ωραία αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή Ανάπτυξη θα συνεχίσει την συνεδρίασή τη ε, στο ε, PHS 4.